Θέλετε Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε. Ελπίζω να περάσετε όλοι καλά. Λίγες βέβαια διακοπές, αλλά ελπίζω να περάσετε καλά. Λοιπόν, μετά το Πάσχα. Λοιπόν, τα ξαναλέμε, καλωσορίστε στο Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα έχουμε το ένα που είναι η έγκριση μερική διάταξης. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάτι να πείτε. Αν όχι, θεωρούμε ότι εγκρίθηκε. Και επίσης σας λέω ότι ε, θα μεταδίδεται και ζωντανά από την ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου η συνεδρίασή μας. Θέμα 2. Η έγκριση των πρακτικών συνεδρίασης 23 Φεβρουαρίου 2010. Εάν ε, μέχρι αύριο το τελειώσει η συνεδρίασή μα δεν έχετε καμία αντίρρηση, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίθηκαν. Τρίτο σημείο, ανακοινώσει τον Προέδρο. Δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή να σας πω. Οπότε περνάμε ήδη στην ψηφοφορία. Ελπίζω όλοι να φέρατε ε, ε, τις κάρτες σας, το, όπως ενημερώσαμε επανειλημμένα. Και ξεκινάμε πρώτα απ' όλα. Τι γίνεται, λέει ο πρόεδρος. Δεν τελείωσα. Μα δεν τελείωσα. <laughs> Περιμένετε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, περνάμε στην έγκριση του προγράμματος τεκμηρίωσης αλληλευμάτων για τον ερυθρό τόνο με εισηγητή τον κύριο Ρωμέβα. Και όπως είχαμε πει, η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα. Κυρία Λοβίν, έχετε ζητήσει το λόγο. Yes, I wonder if we could do the... Ναι. Μήπως θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε διανατάσεως ε, ε, της χειρός. Φαίνεται ότι την έχασα την κάρτα, μάλλον την ξέχασα στο Στρασβούργο. Sí, eh, eh. Ναι, ναι. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Βεβαίω μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο της, ε, της κάρτας σας. Στείλτε κάποιον να ζητήσει. Εντάξει, τη χάσατε στο Στρασβούργο, το καταλαβαίνω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πάρετε μία εδώ σήμερα. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, θα προτιμούσα. Κύριε Ρωμέβα, έχετε το λόγο, αν θέλετε κάτι κάποια σχόλια. Eh, Πρώτα απ' όλα, ε, κάνω κάποια σύντομα σχόλια για να δούμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με την ψηφοφορία. Γιατί έχει κάποιε ιδιαιτερότητε η ψηφοφορία. Είναι καθαρά τεχνική φύσεω, γιατί εδώ πρόκειται ε, για ένα έγγραφο το οποίο ήδη έχει εγκριθεί στην ICAT στα πλαίσια του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, αλλά εδώ υπάρχουν ορισμένα συστήματα τα οποία είναι σημαντικά. Πρώτο, ε, ε, για πρώτη φορά εδώ στην Επιτροπή μας ε, ε, ακολουθούμε το νέο σύστημα. Οπότε πρέπει να ε, συμφωνήσουμε και σε κάποια μέτρα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος. Με αυτή την έννοια έχουμε μια σειρά τροπολογίες που τι αναλύσαμε μέχρι τελευταία στιγμή για να δούμε κατά πόσο πράγματι ήταν σκόπιμε ή όχι. Οι 1 έω 5 οι τροπολογίε αυτέ που έχουν ε, να κάνουν ακριβώ με τον ρυθμό του νομοθετικού πλαισίου. Επίση, έχουμε μια. Ε, οι νομικέ υπηρεσίε μα ε, έκαναν την εξή σύσταση. Το περιεχόμενο αυτών των τροπολογιών που αναφέρεται στα τμήματα της συνθήκης που θα πρέπει να εφαρμοστούν θα, ε, εφαρμόζεται στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Άρα δεν, ε, ε, δεν υπάρχει όμως και λόγος να μην συμπεριληφθούν στην έκθεση. Ταυτόχρονα σας πω ότι η σύσταση των νομικών υπηρεσιών είναι να επαναλάβουμε τις τροπολογίες από 1 ως Και εγώ προσωπικά βλέπω το θέμα ω εξή, ω συζητητής. Δεδομένου ότι δεν παρεμβαίνω στη διαδικασία, νομίζω ότι δεν ε, υπάρχει πρόβλημα να τι διατηρήσουμε. Είναι παραθέσεις που νομίζω ήταν χρήσιμε και για το μέλλον. Γι' αυτό λέω να τι κρατήσουμε τι τροπολογίε αυτέ. Εφόσον έχω ε, ε, ε, ε ω συγκριτή τη δυνατότητα αυτή. Έχουμε αυτή την υπόδειξη των νομικών υπηρεσιών να μην συμπεριληφθούν, αλλά εγώ λέω να συμπεριληφθούν. Δεύτερον, πολύ, πολύ περιληπτικά. Έχουμε μία προφορική τροπολογία που παρουσιάστηκε και βρίσκεται στο τέλος του καταλόγου ψηφοφορίας. Στην ουσία ε, πρόκειται για ένα γλωσσικό ζήτημα. Στο αρχικό έγγραφο το οποίο παρουσιάσαμε και που ήταν στα αγγλικά, η λέξη farm που θα έπρεπε να υπάρχει έγινε for. Γι' αυτό ορισμένες ε, μεταφράσεις ήταν λάθος. Οπότε η προφορική τροπολογία αφορά το πρωτότυπο, το αγγλικό. Εκεί όπου αναφέρεται form πρέπει να λέει farm. Τυπογραφικό λάθος. Και από εκεί θα ακολουθήσουν και διορθώσεις άλλες μεταφράσεις. Κατά τα άλλα δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να ευχαριστήσω τις συγκίτρες και τους συγκητές στους ε, Κιώδης, γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο, ε, στο οποίο υπήρξε αρκετά μεγάλο βαθμό συνένεση. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Αν συμφωνείτε πρώτα, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες αυτές και πάμε να ψηφίσουμε. Πρώτα απ' όλα ψηφίζουμε την 69. Άρχεται ψηφοφορία. Έληξε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 του συγκητή άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 του εισηγητή. Άρχεται. Έληξε. Εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτει η 9, 70 και 71 που αποσύρθηκε. Τροπολογία 10. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 72 αποσύρθηκε. 73. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 74. Άρχη. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 75. Αρχή. Σε la Πέρας. Εγκρίνεται. 11. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 12 αποσύρθηκε. 76 τώρα. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 13. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 14 αποσύρθηκε. Η 77 τώρα αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 15 αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 16 αρχή. Τέλος. Εγκρίνεται. Η 17 αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. Η 18 αποσύρθηκε και πάμε στην 78 αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 19 αρχή. Τέλος. Εγκρίνεται. 20 αρχή τέλος εγκρίθηκε 21 αρχή λήξη εγκρίθηκε 22 αρχή 22 αρχή. Λήξη. Εγκρίθηκε. 23 αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. 24 αρχή, λήξη, εγκρίνεται. Τροπολογία 25, αρχή, λήξη, εγκρίνεται. 26, αρχή, Λήξη. Εγκρίνεται. 79 δεν ψηφίζεται, είναι γλωσσική φύσεως θέμα. 27 λοιπόν του εισηγητή που είναι ταυτόσιμη με την 80. Αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. Στη συνέχεια πάμε στην 28 αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. 81, γλωσσική φύσεως, δεν ψηφίστε. 83, του εισηγητή αρχή. Τέλος. Εγκρίνεται. Η 82 δεν την ψηφίσουμε, ούτε το 4. Πάμε λοιπόν στην 29. Αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. 30 του εισηγητή αρχή. Εγκρίνεται. Οι 31, 32 και 85 αποσύρθηκαν, οπότε πάμε στη 33. Αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. 34 του εισηγητή. Αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. 35 αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. 36 του εισηγητή αρχή. Λήξη. Απροβάδα. Εγκρίνεται 86, δεν ψηφίζουμε. 37 αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. 38 αποσύρθηκε. 39. Αρχή. Πέρασε. Εγκρίνεται. 40 αποσύρθηκε. 87. Αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. Η 88 καταπίπτει. 89 αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτει η 90. Και πάμε στην 91 για την οποία ζητήθηκε ε, ψήφο σε δύο τμήματα ολόκληρο το κείμενο ε, έξω από την τελευταία φράση της παραγράφου 1. Ολόκληρο το κείμενο εκτός από αυτή την πρόταση. Ψηφίζουμε. Λήξη. Εγκρίνεται. Τώρα, την τελευταία φράση της παραγράφου 1. Αρχή της ψηφοφορίας. Πέρας. Επίσης εγκρίνεται. 92. Και εδώ έχει ζητηθεί χωριστή ψήφος. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ολόκληρο το κείμενο εκτός από το τελευταίο τμήμα της παραγράφου 2. Αρχή για αυτό το πρώτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα υποβάλλει προσφορία το τελευταίο τμήμα της παραγράφου 2. Αρχή. Λήξη. Απορρίπτεται. 14 προς 6. 93 του εισηγητή. Αρχή. Πέρασε. Εγκρίνεται. 41 του εισηγητή. Αρχή. Λήξη. Επίσης εγκρίνεται. Καταπίπτουν 99, 100, 94, 95, 96, 97-98 και πάμε στην 44. Αρχή για τη 44. Λήξη. Απορρίπτεται. Ναι, 13 ψηφοφορίες. Με 13 ψήφους, συγγνώμη, 102 αποσύρθηκε, και τώρα υποβάλλω στη ψηφοφορία την προφορική τροπολογία 2 του κύριου Μιλάνα που βρίσκεται στο παράρτημα η τροπολογία του κυρίου Μιλάνα. Ελπίζω να μην διαφωνεί με αυτή την προφορική τροπολογία κάποιος, με τη συμπερίληψή της δηλαδή, άρχεται ψηφοφορία για την προφορική τροπολογία 2. Λίγη. εγκρίνεται. 101 καταπίπτει, 42 αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 43 αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. 45 του εισηγητή. Αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. 46 του εισηγητή τώρα. Αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. 104 δεν την ψηφίζουμε. Ούτε και την 103. 105 αποσύρθηκε. 106 δεν ψηφίζεται. 47. Τροπολογία 47. Αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτει 7 και φτάνουμε 48. Τροπολογία 48 του συγκητή αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49 του εισηγητή, αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται καταπίπτει, επομένως η 108. Και φτάνουμε στην 50. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 109 και υποβάλλω σε ψηφοφορία την 51. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει η 110. Και πάμε στην 52 του εισηγητή. Εδώ έχουμε σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της 52 αρχή λήξη. Εγκρίνεται. Δεύτερο σκέλος. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 111 δεν ψηφίσουμε. 112 δεν ψηφίζουμε. 113 καταπίπτει γιατί έγινε δεκτή 52. Και η 110 καταπίπτει. 115 και αυτή καταπίπτει και η 116. 117, 118, όλες αυτές καταπίπτουν, 53 πάμε, άρχεται. Αρχίζουμε, ε, άρχεται η ψηφορία για το 53. Σε cierra la votación. Λήξη. Εκρίνεται. 120 είναι ταυτόσιμη ε, δεν ψηφίζουμε, 139 δεν την ψηφίζουμε, ούτε 121. Πάμε στην 54. Άρχεται Σε φιέρα, Λίγη. Εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτει 122. Πάμε στην 55. 55. 55 αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 56 αποσύρεται και πάμε στην 123 του εισηγητή. 123 άρχεται η ψηφορία. Λίγη. Απορρίπτεται με 12 κατά και μόλις 9 υπέρ. 123 απορρίφθηκε. Πάμε στην 124. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. 125 δεν Πάμε στην 57. Αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. 58 του εισηγητή αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. 59, τώρα, ναι, 59. Αρχή. Πέρας. Εγκρίνεται. Εξήντα του εισηγητή αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. 61 του εισηγητή αρχή. Λήξη. εγκρίνεται. 62 του εισηγητή αρχή λήξη. Εγκρίνεται. 63 του εισηγητή αρχή λήξη. Εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν, όπως συμφωνήσαμε με τον εισηγητή, 1, 2, 3, 4, που αναφέρονται ότι έχουν αποσυρθεί, αλλά πήραμε την απόφαση να τις φύσουμε. Λοιπόν, 1, αρχή, λίγη. Δύο, του εισηγητή αρχή λήξη. Εγκρίνεται. Τρία, του εισηγητή αρχή Λήξη. Εγκρίνεται. Τέσσερα του εισηγητή. Λήξη. Εγκρίνεται. Πέντε. Αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. 6. Αποσύρθηκε. 65. Αρχή. Λήξη. 66 Καταπίπτη. 7 του εισηγητή. Θα την υποβάλλω για ψηφοφορία. 7. Λίγη. Απορρίπτεται. 67 αποσύρθηκε. 68 του συγκητή αρχή. Λήξη. Εγκρίνεται. ε, πρόταση Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε αρχή πέρας εγκρίθηκε με 20 ψήφους και μία αποχή και θέτω σε ψηφοφορία το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Αρχή πέρας εγκρίθηκε με 19 υπέρ και μία αποχή. Συγχαρητήρια για το αποτέλεσμα της προφορίας. Συγχαρητήρια κύριε Ρωμέβα. A continuación pasamos a votar. Και τώρα στη συνέχεια θα ψηφίσουμε το επόμενο σημείο, το υπαρθμό 5 της διατάξεως, το οποίο αφορά την έκθεση για την ε, εφαρμογή της ε, νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ε, την διάσωση της βιοπικιλότητας. Ο δε εισηγητής ή εισηγήτρια μόνο η η κυρία Ισαμπέλα Λέβιν, στην οποία θα δώσουμε ευθύ αμέσω το λόγο για να θέλει κάτι να μας πει πριν να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Θέλετε αλλιώς να ψηφίσουμε. Thank you very much. Uh, I would like to make an oral amendment on Έχω μια προφορική τροπολογία στον Θεό Τροπολογία υπαριθμών 8 για την παράγραφο 7, λέει η κυρία Λέβιν. Θα ήθελα να ψευστεί χωρικά, χωριστά η τροπολογία ε, και να ενταχθεί στο κείμενο ως μια χωριστή παράγραφος και να λέει περιττέρω ε, περαιτέρω σημειώνουμε ότι έχουμε αυτέ τι διαφορετικέ συνθήκε που αφορούν τι ε, θάλασσε γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ω Παρχέλκο και Βαρκελόνη, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πλαίσιο για την προστασία των θαλασσίων οικοσυστημάτων. Διαβάζει γρήγορα η συγκεντρική. Και τώρα λέει πρώτα, προχωράμε στην ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση τη κυρία Λέβιν. Πρώτα-πρώτα, έχουμε την τροπολογία υπαριθμών 1. Ψηφίζουμε. Se cierra la votación. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 2. Ψηφίζουμε. Se cierra la votación. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 4 της ηγητρίας. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. τη συνέχεια με την υπαριθμόν 5. Ε, Εδώ έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα της ε, ε διατάξεις. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται και αυτό το τμήμα της τροπολογίας, αριθμών 6 τώρα, ψηφίζουμε. Πέρας. Αγκρίνεται. Περιθμόν 7. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία περιθμόν 8. Και εδώ έχουμε μια προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Και είπαμε το τελευταίο κομμάτι εδώ πέρα να γίνει μια καινούργια παράγραφος, αλλά θα πρέπει να γίνει χωριστή ψηφοφορία. Έχουμε την αρχική ε, παράγραφο επί της οποίας έχουμε το, την πετροπολογία του κυρίου Αρσένη. Να το, το διαβάσουμε, όχι. Να ψηφίσουμε όπως είπε η συγγήτρια. Η τροπολογία του κυρίου Αρσένη θα γίνει χωριστή παράγραφος. Και τώρα ψηφίζουμε την τροπολογία Αρσένη ως χωριστή αυτόνομη αυτοτελή παράγραφο και ψηφίζουμε τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται 12-9. Και εδώ το τροπολογία υπαριθμών 9, η οποία είναι συμβατή με την υπαριθμών 8, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Το βόλιο υπαριθμών 10. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 11 της εισηγήτρες. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται με 12. Ε, ναι, υπαριθμών 12 τώρα της εισηγήτριας. Ψηφίζουμε. Se cierra Πέρασε. νούμερο 3. Εγκρίνεται και πάμε στην υπαρμόν 13 του κυριου ρασενε Ρασένη. Ψηφίζουμε. Πέρασε. 12-9. Εγκρίνεται. Υπαρμόν 14. Ψηφίζουμε. δεν Εγκρίνεται. Τροπολή υπερθυμών. 15. Κάντικ. Ψηφίζουμε. δεν Εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε την αριθμό λοιπόν, 16 του κυρίου Αρσένη. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα η υπαριθμόν 17 του κυρίου Αρσένη με χρωστή ψηφοφορία το πρώτο τμήμα της 17. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και τώρα το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 17. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 14, 7 απορρίπτεται. 18 του κύριου Αρσένη, ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε το κειμένο που τροποποιήθηκε. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. ένα. Συγχαρητήρια κυρία Λέβη. Και τώρα, είμαστε στο σημείο παριθμών 6 της σημερινής διατάξεως, όμως δεν είναι εδώ ο κύριος Σαντινό. Δεν ξέρω αν το αναβάλουμε για αύριο. Άρα, εγώ να κάνω την παρουσίαση. Ο κύριος Αντινόρα δυστυχώς δεν είναι εδώ. Τα ξέρει καλύτερα από μένα. Πάντως θα ήθελα να τον ευχαριστήσω. Για την καλοσύνη που είχε να οργανώσει αυτή την αποστολή για όλους εμάς που συμμετέσχαμε σε εκείνη την αποστολή. Βέβαια δεν είμαστε και τόσο πολλοί από το έλεγχο για λόγους που δεν μπορώ να σας πω, αλλά πάντως ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση εκείνη. γραμματεία μου λέει πάντως ότι αύριο πρόκειται να διανεμηθεί το κείμενο. Πρόκειται για αυτή την αποστολή επομένως στη Σικελία, 29 με 31 Πέμπτου. Πήγαμε σε εκείνη την περιοχή ε, της Σικελίας ε, που είναι κατεξοχήν ε, περιοχή της Ιταλίας που ασχολείται με το ψάρμα. Και είναι δηλαδή το, το μπάλο συγκεκριμένα, ματσάρα δελμπάλο κάπως έτσι, είναι ε, το πιο σημαντικό λιμάνι για αλία στη χώρα. Όσον αφορά το Ξηφία και τον κόκκινο τόνο. Επίσης, είχα μια συνάντηση με το ε, Συμβούλιο για την Έρευνα της χώρας, αλλά και και τον Στιγαλιστικό φορέα της Σικελίας για την ελία, Όπως φαντάζεστε, τα βασικά σημεία ήταν το τι θα γίνει με τα τεχνικά μέτρα για τη Μεσόγειο και το σχετικό κανονισμό. Είναι ένας κανονισμός που ε, εισάγει κάποιες παρεκκλήσεις και τέλη Μαΐου αρχίζει να τίθεται σε ισχύ και έχουμε το άρθρο 6 το οποίο αφορά κάποια σημεία ως προς το βάθος που καθορίζονται για την αλία αλλά και κάποιο μέγεθος ψαριών. Esto medidas técnicas es un tema importante y aquí hubo, se cuestionó por algunos diputados, por algunos, mucha parte del sector que se debería pedir και το μέγεθος των δικτυών για το σχετικό ψάρεμα. Τώρα το αν θα αναβληθεί όχι θέση του κανονισμού είναι κάτι που δεν μας βρίσκει όλους σύμφωνος. Και πάντως ελπίζουμε ότι θα υπάρχει αρκετό χρονικό περιθώριο να προετοιμαστούν όλοι με εξωτορχίζει να ισχύει ο κανονισμός. Υπάρχουν κάποια θέματα λοιπόν που και είναι τη Μεσογείου όσον αφορά κάποιες διακρίσεις που γίνονται, ε, κάτι το οποίο επίσης αφορά και τον Ιταλικό αλληλευτικό στόλο, διεθνείς διακρίσεις σε σχέση με τους γείτονες από την Βόρεια Αφρική. Καταβάλλονται προσπάθειες από την Κομισιόν, τόσο ώστε να υπάρξει εναρμόνιση, τουλάχιστον όσον αφορά τα πιο σημαντικά νομοθετήματα. Ε, αυτό γίνεται μέσω του Συμβουλίου, γίνεται μέσω της ΕΚΑΤ και, και με κάποιες άλλες, ε, με φορείς για να έχουμε καλύτερη εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας για την Μεσόγειο. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα χωρικά ύδατα Τινησίας, Λιβύης και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν διάφορες προστριβές με τη Λιβύη. Είναι τα βασικά προβλήματα αυτά βασικές διεκδικήσεις που προβλήθηκαν κατά τη συνάντηση αυτή στην Σικελία. Και είπαμε πολύ ενδιαφέρουσε επαφέ αυτές για όλους εμάς που ασχολούμαστε και ξέρουμε τα θέματα. Επίσης, Καταλαβαίνετε ότι περάσαμε καλά, γιατί η Σικελία έχει καλή κουζίνα, βάλαμε και κανένα κιλάκι, αλλά οπωσδήποτε και ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός, οπότε ήταν πάρα πολύ θετικό το ότι έγινε αυτή η επαφή λοιπόν από αυτές τις συνθήκες με το αναλυτικό κλάδο στην Σικηλία. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι να σας εξηγήσω. ή Ιδάλλως, σταματάμε εδώ και αύριο αν θέλει ο κύριος ε, αν ώρα μπορεί να μας πει κάτι παραπάνω. Εσείς κύριε Γαντέκ που και εσείς ήσασταν εκεί τι λέτε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω απλά και μόνο ότι αν δεν είχαμε όλοι πιστεί για την ανάγκη περιφερειοποίηση στα πλαίσια της μεταρρύθμισης κοινή ελληνικής πολιτικής, ε, καταλαβαίνετε ότι ε, πιστήκαμε λίγο περισσότερο με, το, με αυτή την επίσκεψη στη Κελία. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πατρά. Ε, ε, ε, Κοιτάξτε, η Πρόεδρος ήδη αναφέρθηκε στο βασικό πρόβλημα το οποίο ε, συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στη Σικελία ε, και αναφέρομαι στο γεγονός ότι η Μεσόγειος ε, αντιμετωπίζει, είναι μάλλον αντικείμενο αλίας από πολλές χώρες. Ορισμένες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν είναι όλες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί πρόβλημα γιατί από τη μια έχουμε τις, ε, Ευρωπαϊ... τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να ε, συμμορφούνται με πιο πολύ πιο αυστηρούς κανόνες από ό,τι οι υπόλοιποι. Ε, έχουμε την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική έτσι ώστε να πετύχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση της αλίας και στη Μεσόγειο. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω και την Πρόεδρο και την Επιτροπή γενικότερα. Μήπως λοιπόν δεν θα έπρεπε ακριβώς ευκαιρία αυτή της επίσκεψης στη Σικελία δεν θα έπρεπε να υπάρξει ένα έγγραφο μια επιστολή αν θέλετε, όπου να τονίσουμε αυτή την ιδέα. Μια, μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Μια πολιτική που θα μπορέσει να μας δώσει την εγγύηση για ε, μια ισότιμη κατάσταση στη Μεσόγειο και για ίσες ευκαιρίες αλίας. Γιατί αν εμείς δεν θέσουμε αυτό το στόχο της ε, από κοινού διαχείρισης των πόρων στη Μεσόγειο, τότε οι παράκτιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρίσκονται όλο και σε πιο μειονεκτική θέση. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε εσείς, πάντως και εγώ μπορώ να σας πω ότι ε, αυτή η επίσκεψη ε, ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Ε, ε, ήταν εντατικό το πρόγραμμα, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, είχαμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες επαφές και πρέπει να σας πω ότι οι επαφές αυτές έγιναν μέσα σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα με, τους, με τον τοπικό πληθυσμό, με τους αλληλείς της περιοχής και με τους συναδέλφους. Δηλαδή όλοι είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε μια ατμόσφαιρα λιγότερο επίσημη θα έλεγα, αλλά πολύ φιλική. Ο κύριος Αντινόρο βεβαίω είναι ο εισηγητή για την ε, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στη Μεσόγειο. Ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με το θέμα αυτό, τα ξέρει ο κύριος Αντινόρο και είναι και από τη Σικελία, άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ο ιδανικός άνθρωπος. Πάντως, ε, ε, οι περιφερειακές οργανώσει οργανώσεις είναι τα κατάλληλα φόρα. Ε, για αυτά τα μέτρα τη ολοκληρωμένη πολιτική. Και βεβαίως ε, πρέπει να προχωρήσουμε την κατεύθυνση αυτή τη ολοκληρωμένη πολιτική. Και σα το λέω, ο κύριο Αντινόρ είναι για αυτή την πολιτική στη Μεσόγειο, οπότε πρέπει να καταβάλει μια προσπάθεια και να μα παρουσιάσει ένα έγγραφο το οποίο ε, να καλύψει ανάγκε μόνο τη Σικελία αλλά και των υπόλοιπων περιοχών τη Μεσογείου. Ωραία. Και πάμε στο επόμενο θέμα τη ημερήσια διάταξη που είναι η νέα όφηση στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια που όλοι ξέρουμε ότι είναι εισηγητής ο κύριος Μιλάνα. Να πω ότι αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Ο κύριος Μιλάνα ήδη έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο έκθεσης, το οποίο το έχετε πάρει στις γλώσσες σας. Και καταρχήν ε, η ψηφοφορία προβλέπεται για τις 4 Μαΐου. Να δώσουμε όμως το λόγο στον κύριο Μιλάνα για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Και στη συνέχεια θα έχουν το λόγο τα μέλη της Επιτροπής. Έχετε το λόγο κύριε Μιλάνα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο γιατί το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Κοιτάξτε, ε, η αρχική αυτή θέση στη γνωμοδότηση που βεβαιώθηκε και μέσα από τις συζητήσεις που είχαμε στο πλαίσιο της Επιτροπής ε, της δικής μας αλλά και με τη δημόσια ακρόαση και με ορισμένα σεμινάρια που έγιναν ε, και σε παιδομάδων και στις συζητήσεις που έγιναν με τους σκιώδεις ηγητές και ε, στη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα αυτά επιβεβαίωσαν την αρχική θέση. Βεβαίω, έχουμε καθυστερήσει το συγκεκριμένο τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ανακοίνωση του 2002 δεν έδωσε τις ε, κατάλληλες απαντήσεις ε, έτσι ώστε ε, να αντιμετωπίσουμε συνολικά το σύστημα αυτό. Η καθυστέρηση σήμερα οδήγησε σε μεγάλη απόσταση και καθυστέρηση της Ευρώπης απέναντι στις υπόλοιπες χώρες όσον αφορά και το αριθμό ανάπτυξης του τομέα αυτού. Πάντως, εδώ στη γνωμοδότηση επαναπροτείνουμε μία σειρά αποζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και που αφορούν ακριβώς το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα, αυτή τη νέα φάση ε, για την προοπτική ανακοίνωση τη Επιτροπής, μην το ξεχνάμε. Και η γνωμοδότηση απαντά στην ανακοίνωση αυτή, λέγοντας ότι πρέπει να βάλουμε τάξη ε, στις, ε, στις διάφορες, στα διάφορα νομοθετικά μέσα τα που υπάρχουν και κανονιστικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητάμε λοιπόν να υπάρξει ένας ενιαίος κανονισμός. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα πρέπει να μιλήσουμε ε, για τον κανονισμό αυτή τη στιγμή και να το γράψουμε τώρα, αλλά να μιλήσουμε για την ανάγκη που υπάρχει να υπάρξει αυτό ο ενιαίο κανονισμό. Και αν θέλουμε να δώσουμε μια θετική όφηση, αυτό άλλωστε αναφέρει και η ανακοίνωση, στην βιώσιμη και αηφόρο ευρωτοκαλλιέργεια, τονίζω αυτό το αηφόρο, ε, θα πρέπει να δημιουργηθεί, να δούμε και την, και την, και ε, δημιουργία ενό ειδικού ταμείου. Ε, είτε στα πλαίσια του Ταμείου της Κοινής Ελευθερικής Πολιτικής και φαίνεται ότι αυτό επικρατεί ως άποψη, και στη συνέχεια να σας πω ότι ε, λέμε ε, πιο συγκεκριμένα τι θα πρέπει να περιέχει αυτός ο κανονισμός. Δηλαδή, πέραν ε, της καθαρά μεθολογικής πτυχής, θέλουμε να δούμε και ποιοτική άποψη, το πώς μπορούμε να εισάγουμε στοιχεία τα οποία θα μας οδηγήσουν ε, σε μια κατάσταση όπου θα μπορέσει να αναπνεύσει ο τομέας, με δύο λόγια. Ε, εδώ αναφέρομαι τα θέματα που έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική επίπτωση αυτών των παρεμβάσεων ε, στον τομέα και θεωρούμε ότι είναι στρατηγική σημασίας ε, η εισαγωγή μια έννοια που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε θαλάσσια χωροταξία και σε επιμέρους περιφέρειες, άρα που θα μπορούσαν να λάβουν τα κράτη. Και όλα αυτά θα αποτελέσουν ένα το οποίο θα μα βοηθήσει να λύσουμε συνολικά το πρόβλημα. Το πρόβλημα τη συμβατότητας των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργεια ε, με τους άλλους παραγωγικούς τομείς, ε, όπως για παράδειγμα ο τουρισμός. Επίσης, τις να δούμε τις επιπτώσεις σε περιοχές όπου θα μπορούσαμε να έχουμε ε, μία ε, παραγωγική δραστηριότητα που να συμβιώνει αρμονικά με τις άλλες δραστηριότητες. Ε, και εδώ να δούμε και το θέμα της υδατοκαλλιέργειας offshore, στην οποία επίσης αποδίδεται στρατηγικός χαρακτήρας. Το έγγραφο το οποίο έχετε μπροστά σας προτείνει διάφορες πολιτικές επιβεβαιώνει την άποψη ότι η δετοκαλλιέργεια δεν είναι ενιαία. Έχουμε ε, την υδατοκαλλιέργεια ε, στα, στο, στα, στο γλυκό νερό, ε, στα, στα θαλάσσια ύδατα. Έχουμε διάφορες μορφές και ο καθένας από αυτούς τους τομείς ε, είναι διαφορετικός. Και ακριβώς εδώ ο κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει μία σειρά από συγκεκριμένα στοιχεία έναντι αυτών των διάφορων μορφών υδατοκαλλιέργειας. Σε τελευταία ανάλυση, το προϊόν ε, ε της στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, αντιμετωπίζει πρόβλημα ανταγωνισμού. Πρόβλημα ανταγωνισμού που προέρχεται από τις εισαγωγές, γιατί κοιτάξτε ο τομέας αναπτύχθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμείς τα τελευταία χρόνια ε, είχαμε ανάπτυξη λίγο πάνω από το 1%. Ε, όμως, ε, στον υπόλοιπο κόσμο όμω υπήρξε ανάπτυξη κατά 6-7%. Άρα καλύφθηκαν οι ανάγκε, αλλά μέσα των εισαγωγών. Το έγγραφο λοιπόν παραπέμπει στην ανάγκη να υπάρξει περισσότερη ρύθμιση σε συνολικό επίπεδο, χωρίς βεβαίω να είμαστε πρόστα, να ακολουθήσουμε πρακτικές προστατευτισμού, αλλά να εξετάσουμε και το θέμα των εισαγωγών. Ε, όσον αφορά το θέμα αυτό, να σα το πω ότι υπάρχει και μια γνωμοδότηση τη Επιτροπή. ο συνάδελφο ε, κατά είναι και αφορά το σύνολο των εισαγωγών στον τομέα της αλίας προς την Ευρώπη. Πάντως στην περίπτωση της ιδετοκαλλιέργειας ε, ε, είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα, σας το ξαναλέω. Εμείς 1,2 εκατομμύρια τόνους ε, προϊόντων υδατοκαλλιέργειας παράγουμε το χρόνο και όμως η κατανάλωση ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Από τη μια λοιπόν θέλουμε περισσότερες εγγυήσεις για τα εισαγόμενα προϊόντα και από την άλλη να δούμε την ανταγωνιστικότητα. Ε, δεν μπορούμε βέβαια να μειώσουμε το κόστος και να έχουμε μόνιμες ενισχύσεις. Δεν μπορούμε διαρκώς να ε, επιχορηγούμε τον τομέα. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε το θέμα της ποιότητας. Και το, τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κανόνες ε, που θα καθοριστούν ε, πιο αυστηρά και πιο συγκεκριμένα από τον κανονισμό θα δώσει ένα πλεονέκτημα στο ευρωπαϊκό προϊόν έναντι του εισαγόμενου. για τα οποία, για τα εισαγόμενα προϊόντα πολλές φορές δεν ξέρουμε πολλά. κοιτάξτε, ε, ε, όσον αφορά το πενγκάς αυτό ε, το, το, συγκεκριμένο προϊόν, εξακολουθούμε όλοι να ε, καταναλώνουμε το ψάρι αυτό και δεν ξέρουμε τι σχήμα έχει. Ε, άρα λοιπόν, εντάξει, αστε, αστειευόμαστε, αλλά θα πρέπει να δούμε τώρα τι ακριβώς γίνεται και κανένας δεν ξέρει, δεν έχει κανένα στοιχείο για το θέμα αυτό. καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά για την προστασία του καταναλωτή υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο παραμένει ανοιχτό και το οποίο θα πρέπει να το δούμε και στα πλαίσια του συγκεκριμένου κανονισμού στα οποίο αναφέρομαι και που αναφέρεται στη στήριξη τη τεχνολογική καινοτομία και στην επιστημονική έρευνα. Και γιατί κάνω διάκριση στα δύο ζητήματα. Από τη μια, η επιστημονική έρευνα είναι αυτή που μα βοηθά. Και πρέπει να σα πω ότι ε, ε, πρόσφατα ε, και μάλιστα θα μπορούσα και εγώ να προτείνω ε, τροπολογία, γιατί πρόσφατα έμαθα πολλά στοιχεία και μάλιστα μόλι είχα ολοκληρώσει την εργασία μου. Ε, για παράδειγμα, στον τομέα των ζωοτροφών, που είναι ένα τομέα στον οποίο είχαμε πολλέ διαφορέ και, και πολλέ συζητήσει. Λοιπόν, η, η, έρευνα έχει προχωρήσει πολύ προ από εμά, επιστημονική. Με την έννοια ότι αυτά που για μας ήταν στόχοι εντό εισαγωγικών στρατηγικού ή πολιτικού χαρακτήρα. Δηλαδή η μεγαλύτερη χρήση φυτικών πρωτεϊνών έναντι των ζωικών. Ε, να βγούμε δηλαδή από την παλιά κατάσταση όπου τα, ε, τα ψάρια καταναλώνουν ψάρια, αν θέλετε. Ε, λοιπόν, εδώ οι επιστήμονε έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο και δίνουν την έμφαση ακριβώ στα ζητήματα τα οποία συνδέονται με την ποιότητα των ζωοτροφών, των ε, ηχθειοτροφών, αν θέλετε τα περίφημα, τα περίφημα ζητήματα ε, που έχουν να κάνουν με την προστασία των ιδιωτήτων των, ε, των ηχθείων. Παράδειγμα, μείωση της χολυστερίνης, θέμα στο οποίο δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και οι καταναλωτές. Ε, λοιπόν, εδώ η έρευνα ε, έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο, όπως σας είπα, και αναφέρεται συγκεκριμένα και με αποτελεσματικό τρόπο στα ζητήματα αυτά τόσο όσον αφορά δηλαδή στη διατήρηση των ποιοτικών προτύπων, αλλά και κυρίως από την άποψη ε, του, της αναλογίας ε, των φυτικών πρωτεϊνών έναντι των ζωικών. Έχουν προχωρήσει λοιπόν πολύ προσφορά από ό,τι και εμείς τα προσδοκούσαμε. Βεβαίω το ζήτημα αυτό είναι ανοιχτό, γιατί έχει να κάνει και με την ανάκτηση ε, ε πολλών ε, θεακών πόρων, ε, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή, ε, παραγωγή αλεύρων ε, ε, και ελαίων, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία εντάσσονται σε αυτό το σύστημα όπου θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για έλλειψη ισορροπίας σε αυτή τη διατροφή των ηχθείων. Τώρα, όσον αφορά το τεχνολογικό ζήτημα, ένα είναι το επιστημονικό και όσον αφορά το τεχνολογικό ζήτημα, και εδώ έχουμε μεγάλη πρόοδο. Ε, όσον αφορά τι εγκαταστάσει, για παράδειγμα. Τι σύγχρονε εγκαταστάσει που χρησιμοποιούν ιδιαίτερη τεχνολογία. Για παράδειγμα, με στόχο τη μείωση των ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται και που χάνονται στο νερό, διαλύονται στο νερό. Εδώ αυτό έχει να κάνει με συγκεκριμένη τεχνολογία. Όταν δηλαδή κανείς χρησιμοποιεί τροφές σε μία ε, υδατοκαλλιέργεια, καταλαβαίνετε ότι μέρος της τροφής καταναλώνεται απευθείας από τα ψάρια τα οποία είναι στη θάλασσα, έτσι. Και ένα τμήμα, ακριβώς για, λόγους, για τεχνικούς λόγους, και κάποια καθυστερημένη τεχνολογία, εφαρμογή τη τεχνολογία σε ορισμένε περιπτώσει, κάποια καθυστέρηση που υπάρχει, ε, διασκορπίζεται στη θάλασσα. Ε, αυτό όμω έχει αρνητικέ επιπτώσει και στο περιβάλλον. Γιατί ε, ε έχουμε αυτέ αυτά τα, αυτές τις αντίξωες ε, επιπτώσεις στο, στο θαλάσσιο περιβάλλον. Και εδώ λοιπόν η τεχνολογική έρευνα πέραν της επιστημονικής αποτελεί ένα μέσο το οποίο σίγουρα μπορούμε να το, να το χρησιμοποιήσουμε γιατί μας βοηθά προς την κατεύθυνση αυτή. Ένα άλλο ζήτημα και τελειώνω πολύ σύντομα, αφορά το τέλος του κύκλου αυτού. Δηλαδή πολιτική σήματος στο τέλος της διαδικασίας. Στήριξη λοιπόν πολιτικής ε, σήματων που γίνεται μέσω της ε, πιστοποίησης του προϊόντος, του ελέγχου του κυκλώματος στο σύνολό του και αυτή η πολιτική ε, σήματος και εικόνας έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με το βιομηχανικό ευρωπαϊκό προϊόν και από την άλλη με τα βιολογικά προϊόντα. Ε, και εδώ, ε, παραπέμποντας και σε πρόσφατους κανονισμούς, που ήταν, θα έλεγα, προϊόν ε, προώθησης ε, της ε, βιολογικής γεωργίας και δεν αφορούν συγκεκριμένε δραστηριότητε, αν θέλετε αλλά που όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να το δούμε ε, τι επιπτώσεις έχουν στο συγκεκριμένο τομέα. Η ε, στρατηγική σημασία για μα είναι η διασφάλιση τη υγεία των ηχθείων. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε μια πολιτική για το ευρωπαϊκό σήμα συνολική. Από τη μια λοιπόν έχουμε το, το βιομηχανικό προϊόν, επιτρέψτε μου χρησιμοποιήσω τον όρο αυτό, παρόλο που δεν είναι απόλυτα σωστός, και από την άλλη ε, η βιολογική παραγωγή. Και όλα αυτά σε μια φάση όπου γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά ότι ε, υπάρχει πρόβλημα ελέγχου των αποθεμάτων των ηχθείων που βρίσκονται στη θάλασσα. Αυτό είναι συνολικό ερώτημα. Άρα λοιπόν ε, η υποτίμηση του συγκεκριμένου τομέα είτε μπορεί να μας οδηγήσει ε, σε σημαντική έλλειψη της ζήτησης είτε ε, να δημιουργήσει προβλήματα και σε επίπεδο παραγωγής και απασχόλησης. Να σας, πω, να σας εξηγήσω τι θέλω να πω. Εδώ βλέπουμε συνολικά το μέλλον της αλίας που συνδέεται με μείωση και των απασχολούμενων, έτσι. Κυρίως των απασχολούμενων στον τομέα αυτό. Και αυτό λόγω του τρόπου Ελίας που γίνεται όλο και πιο αποτελεσματικός. Άρα, αν θέλετε, ε, απαιτείται μικρότερος αριθμός εργαζομένων και από την άλλη έχουμε συνολική μείωση των ε, αποθεμάτων των ηχθείων. Μία λοιπόν επαρκής και σωστή πολιτική για την ιδετοκαλλιέργεια θα μπορούσε να βοηθήσει και προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί θα μπορούσε η ιδετοκαλλιέργεια να αποτελέσει το κατεξοχήν μέσο για την ανάπτυξη των θέσεων εργασίας και ίσως και μέσω της ε, ε, προσφυγής σε προγράμματα κατάρτισης, αν θέλετε. Αναδιαμόρφωσης λοιπόν αυτού του εργατικού δυναμικού που ε, το διώχνει, αν θέλετε, την παραδοσιακή αλληλεία και που μπορούμε τώρα να ενσωματώσουμε στα πλαίσια μιας υγιούς και αϊφόρου εξέλιξης ε, της ερωτοκαλλιέργειας. Αυτά ήθελα να πω. Νομίζω ότι συνόψισα πολύ σύντομα αυτά τα οποία έχετε μπροστά σας και γραπτά. 14 Απριλίου νομίζω ότι ορίσαμε για τις ε, τροπολογίες. Εγώ πάντως είμαι διαθέσιμος, είμαι στη διάθεσή σας. Ε, Όποιο συνάδελφος θέλει να συζητήσουμε κάποια στοιχεία και να δούμε τι μπορεί να γίνει με τις τροπολογίες, συνεχίζοντας αυτή την εργασία, ε, την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής και με τους κοιόδους ηγητές και με όλους τους συναδέλφους λοιπόν που θεωρούν σκόπιμο, είμαι στη διάθεσή σας μέχρι την προθεσμία αυτή θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση στι αρχές Μαΐου στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια του Μαΐου ή του Ιούνιου. Ή του Ιουνίου. Είμαι στη διάθεσή σα λοιπόν για περαιτέρω παρατηρήσει και σκέψει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, θα, θέλαμε να, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή για μια εξαιρετική έκθεση. Ε, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε πολλά ζητήματα σας, γιατί ήδη καλύψατε πάρα πολλά από την πλευρά σα, ειδικά για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ε, διασφάλιση του να υπάρχουν τοπικές εκμεταλλεύσεις οι οποίε θα επιβιώσουν και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας και από την πτυχή της πιστοποίησης είναι ε, όλα σημαντικά ζητήματα τα οποία αναφέρεται μέσα σε αυτήν την γνωμοδότηση. Όμω θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή ιδιαίτερα σε ένα ζήτημα που και αυτό το αναφέρατε. Και αυτό είναι το εξή. Η θέσπιση ε, νομοθεσία σε ό,τι αφορά την ευμερία των ζών θα πρέπει να καλύπτουμε και ζητήματα όπως αυτό της ε, πυκνότητας, δηλαδή της συγκέντρωσης των νυχθείων ανά κυβικό μέτρο. Δηλαδή θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη μας τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε τρεφόμενου είδους και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ούτως ώστε να αποφύγουμε να υιοθετήσουμε ορισμένες διατάξεις πολύ πρόωρα, πολύ βιαστικά. Άρα λοιπόν τέτοιου είδου ε, πολύ αυστηρέ ε, διατάξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται στις ε, οργανικέ βιολογικέ δηλαδή. Ηχθειοκαλλιέργειες, ούτω ώστε να μην εντατικοποιηθούν σε ό,τι αφορά δηλαδή το βαθμό εκμετάλλευση σε τέτοιου είδου εκμετάλλευση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Συγχαρητήρια που στον εισηγητή για όσα μα είπε γιατί η έκθεσή του φύγει πολύ σημαντικά ζητήματα και είναι πάρα πολύ σωστό το ότι λέμε θα πρέπει να υπάρχει έτσι ένα πλαίσιο οικονομικό, διοικητικό, νομοθετικό και κάτι που να αφορά την ποιότητα του προϊόντος. Τώρα θέλω να σας πω κάτι όσον αφορά την, ε, την πολιτική της χωροταξίας ας πούμε ε, που παρουσιάζει ενδιαφέρον σαν θέμα γιατί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτή την συμβατότητα της βιώσιμης ικτιοκαλλιέργειας με το δίκτυο Συμφωνώ ότι υπάρχει συμβατότητα, όμως θα πρέπει να κάτσουμε εδώ και να δούμε ότι η πρώτη επιλογή είναι η χώρη προστασίας, όπου θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη υπό ποιες προϋποθέσεις χώρη τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, έχουμε κάποιες μεγάλες ε, νυχτιοκαλλιέργειες ή κάποια εξωτερήκευση όσον αφορά τα φάρμακα, τη, τη διατροφή των ψαριών όπου υπάρχουν και άλλες ε, μεταβλητές. Άρα θα πρέπει εδώ πέρα να διαφοροποιήσουμε το τι λέμε, το τι ζητούμε, για να μην έχουμε κάποιο είδου παραθυράκι για κάποιες τέτοιες χτιοκαλλιέργειες. Όταν να αφορά τις εισαγωγές, οι έλεγχοι και τα μέτρα τα σχετικά παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τι γίνεται να δούμε με τους λιμένες εισαγωγές και εισόδου και να δούμε πώς με κατάλληλους ελέγχους θα έχουμε κάποιες εγγύησης ισότητα μεταχείρισης των προϊόντων των εισαγόμενων με τα δικά μα. Πρόεδρος. Έχω και εγώ κάποιε παρατηρήσεις. Πρώτα πρώτα. Μετά τη του 48 του κανονισμού και λέτε εκεί σε αυτή την, ε, την τελική παράγραφο ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ποιο κανονισμό? όμως. άρα εδώ θα πρέπει να διευκρινίσετε σε ποιον κανονισμό παραπέμπεται. Επίσης, θα ήθελα να δούμε τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ελίας. Κάποιε από τις παρατηρήσεις που αναφέρεται, ας πούμε, στη διάταξη παρτιμών 25, είναι θέματα τα τα καλύπτει τώρα ήδη το Ταμείο Ελίας. Και Τότε που συζητήσαμε τη σχετική έκθεση, ζητήσαμε να καλυφθεί και η καλλιέργεια, γιατί είπαμε δεν θα πρέπει να υπάρχει τέτοιο διαχωρισμό όσον αφορά τις ενισχύσει. για τι ΜΜΕ από τη μία και από την άλλη μεριά για κάποια μεγάλα προγράμματα. ξέρετε και αυτό και για την δική σας έκθεση. Απαιτούνται εδώ σημαντικές ε, επενδύσει, αλλά δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε σε ενισχύσει προ τι να αναζητηθεί από το Συμβούλιο να μας καλύψει και σε αυτό το θέμα που δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Άρα πρέπει να κατεβάσουμε μια, μια σχετική τροπολογία τώρα. Αυτό που ο κύριος Πρασέδο για αυτή την ιτολογική παράγραφο. Βεβαίω και δεν υπάρχει ασυμβατότητα. Νομίζω ότι συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένα το έχει πει για το δίκτυο να Natura δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε το σημείο αυτό, 25. Για αυτά τα προϊόντα ιδιωτοκαλλιέργειας και τις κοινέ οργανώσεις αγορών ότι η Ταμείο Αλίας τι θα πρέπει να καλύψει. Αν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει μια τέτοια πρόβλεψη. Άρα, με κάποιες τοπολογίες να κάτσουμε για να διευκρινίσουμε αυτά τα ζητήματα. Όμως, επί του συνόλου δεν έχω καμία ένσταση. Έχετε το λόγο. Ε, Πατράου. Πατράου. Eh, eh, Ευχαριστώ. Ε, με ευχαριστεί το γεγονό ότι έχει προβλέψει ω ιδέα μέσα στην νομοδότηση ε, ο ζήτης ε, ένα σήμα ποιότητας, ε, ένα είδος σήματος ποιότητας λοιπόν για τα προϊόντα που θα προέρχονται από αυτές τις υδατοκαλλιέργειες και θα ήθελα εδώ να τονίσω το εξής. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα επιμέρου ζητημάτων, ώστε αυτή η πολιτική ποιότητα, αυτή η πολιτική προστασία του καταναλωτή να διαμορφωθεί με τρόπο τέτοιο, έτσι ώστε να μην προκληθεί υπερβολική σύγχυση στους ίδιους τους καταναλωτές. Δηλαδή να μην δημιουργηθεί τελικά μια πληθώρα από τέτοια σήματα ποιότητας. Και θα ήθελα ε, σε σχέση με αυτό το ε, ζήτημα να ε, σας παραβέμψω και στο ζήτημα της πιστοποίησης των υδατοκαλλιεργειών και στον οργανισμό τροφίμων και γεωργίας των ΕΦΕΟ των Ηνωμένων Εθνών ε, έγιναν ε, και κάποιες ε, σχετικές συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο. αναφέρθηκαν εκεί τέσσερις βασικές πτυχές και ίσως θα είχε νόημα να εξετάσουμε λοιπόν εκείνες τις πληροφορίες στο πλαίσιο της εν λόγω έκθεσης. Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες τροποποίησεις αν λάβουμε αυτά τα στοιχεία απόψε. Σα ευχαριστώ. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ άρτη αυτή η έκθεση και θα περιοριστώ επομένω να κάνω κάποια γενικά σχόλια όσον αφορά την νομοτεχνική πλευρά. Ο κύριο ε, Λάνα θέλει να υπάρχει μια τέτοια τομιακή προσέγγιση για την ιχθυοκαλλιέργεια. Ε, μια κάθετη προσέγγιση και έτσι όλες οι διαστάσεις της ηθοκαλλιέργειας να μπουν ε, σε μια εκθεσή όπως ε, τα λέει το σημείο παραγωγός 15 και έτσι να έχουμε και το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος περιβάλλον και ηθοκαλλιέργεια η αμοιβαία επίδραση η καλονταχείριση των ζώων η δημόσια υγεία η χρήση των σχετικών φαρμάκων όσον αφορά την ηχιοκαλλιέργεια, την αχνευσιμότητα, την πιστοποίηση των προϊόντων της ηχιοκαλλιέργειας, την εμπορική πολιτική, όλα αυτά. Τη χωροταξία, τις κρατικές ενισχύσεις, την προσβασιμότητα στην ε, παραλία και στα ιστορικά ύδατα. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι ακριβώς αυτή που σήμερα ήθεστε να ακολουθούμε πολλές νομοτεχνικές Κάθε άλλο όσον αφορά το κοινοτικό δίκαιο τουλάχιστον γιατί πρόκειται για κάποια προσέγγιση που θα πρέπει να την ζυγίσουμε, να την αξιολογήσουμε. Όσον αφορά το δημόσιο δίκαιο. Μάλλον οριζόντια κινούμεθα όσον αφορά τη σχετική νομοθεσία. Αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Οπότε, κατά κλείδι, σα τονίζω ότι στα πλαίσια του προγράμματο εργασία τη 31η Μαρτίου για το 2010 δημοσιεύουμε στο δεύτερο παραρτημά μα μία ενδεικτική λίστα, έναν κατάλογο για τι πρωτοβουλίε τις οποίε δίνουμε προτεραιότητα. Ούτω ώστε να προχωρήσουμε για το 2010 στην υιοθέτηση σχετικών μέτρων και έχουμε και νομοθετικέ προτάσει, ούτω ώστε να υπάρξει μια δέσμη μέτρων για μεταρρύθμιση τη και εκεί να καλύψουμε και την ε, ηχθειοκαλλιέργεια. Επομένως είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό ε, σε σχέση με το πρόγραμμά μας αυτό το οποίο γίνεται τώρα. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Να διευκρινίσω όμως το εξής. Αυτό, αυτή εδώ η γραμμή δεν έχει να κάνει, καμία, ε, δεν έχει να, δεν έχει να κάνει κάτι με το έγγραφο. Ε, είναι λάθος, τυπογραφικό. Μάλιστα, δεν το, δεν το πρόλαβα και δεν το είδα. Δεν έχει να κάνει όμως καμία... Ε, δεν, δεν έχει καμία σχέση. Δεν υπάρχει κανένα άρθρο 48 και κανένας κανονισμός. Πράγματι. Υπάρχει ένα κόμμα. <laughs> Είναι μόνο τυπογραφικό το, έχοντας υπόψη λοιπόν σταματά στο ΦΑΟ και στο μη υπεύθυνη Ελία. Τώρα, ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι πήραν το λόγο, ε, τον πρόεδρο, την πρόεδρο, τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ ε, με όσους τοποθετηθήκατε και να σας πω το εξή. Αυτή τη στιγμή δεν γράφουμε τον κανονισμό, έτσι. Σχολιάζουμε μία ανακοίνωση της Επιτροπής αν ε, γράφαμε τον κανονισμό, θα ήταν τελείως ανεπαρκή η γνωμοδότησή μου, έτσι, αλίμονο. Ε, προς Θεού, εδώ θέλουμε ε, να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα με σοβαρότητα βεβαίως, το τονίζω. Και κάτι άλλο, όσον αφορά το τελευταίο αυτό ζήτημα, το συζητήσαμε με τους υπεύθυνους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμένα δεν με τρομάζει η καινοτομία και όσον αφορά την νομοθετική τεχνική δεν με ενισχύει καθόλου το ζήτημα αυτό και θα μπορούσαμε να προτείνουμε διαφορετικές μεθόδους. Αν θεωρήσουμε ότι ο τομέας ο συγκεκριμένο πρέπει να αναπτυχθεί, τότε γιατί, αν ναι, ε, αν συμφωνούμε, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε και νέε μεθόδου. Σα το λέω ε, με κάθε μετριοφροσύνη ε, προ Θεού. Ε, δεν έχω την πρόθεση να διαταράξω τι διαδικασίε, αλλά σα πω το εξή. Οι μορφέ λήψη απόφαση όταν μιλάμε αυτή τη στιγμή για νομοθετική τεχνική ή για βασικές επιλογές, θα μπορούσαμε να εισάγουμε και το στοιχείο της καινοτομία. Θα το συζητήσουμε. Βεβαίω δεν μπορούμε να έχουμε πρόβλημα με την ε, νομική επιτροπή. Την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θα έχουμε περαιτέρω συζητήσει. Αλλά και εμεί ε, ω Επιτροπή Ελία θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάποια στοιχεία καινοτομία που να μα οδηγούν σε αποτελεσματικότητα. Κατά την άποψή μου, αυτό που ενδιαφέρει ε, είναι το Κοινοβούλιο να λέει σαφώ την άποψή του και να εισάγει στοιχεία τα οποία αντιμετωπίζουν συγκεκριμένε ανάγκε, αν υπάρχουν αυτέ οι ανάγκε, με συγκεκριμένε ε, απαντήσει. Και εφόσον η ανάγκη εντοπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μα έδωσε την ανακοίνωση και ζητήθηκε η γνωμοδότησή μα, ε, σε αυτή την ανάγκη λοιπόν εμεί προσπαθούμε να απαντήσουμε με του όρου αυτού. Επομένω, όλα αυτά τα οποία Ε, και εδώ σας παραπέμπω και στην ε, παρέμβαση της κυρίας Πατράου που είναι πάρα πολύ κέρια. Όταν εγώ μιλώ για πολιτική σήματο, μιλώ για τον ορισμό των χαρακτηριστικών και για τη χρησιμοποίηση του σήματο στα πλαίσια τη κοινοτική λογική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άρα πρέπει να επισέλθουμε στη λογική κοινοτικού σήματο. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, την ιδιωτοκαλλιέργεια μεμονωμένη, αλλά μέσα στα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε τα χαρακτηριστικά τα οποία ε, χρησιμοποιούνται ως επιχείρηματα για να υποστηρίξουν το σήμα θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα, δεν μπορεί να είναι γενικά. Και θεωρώ ότι, σας το λέω καθαρά, ε, ε πέρυσι είχαμε ένα κανονισμό που αφορούσε τη βιολογική δεδοκαλλιέργεια στα πλαίσια μιας συζήτησης επευκαιρία της συζήτησης για την βιολογική γεωργία. Χωρίς το Κοινοβούλιο και βεβαίως ε, ε, και στη δική μας την Επιτροπή ε, να πούμε την άποψή μας. Ε, βεβαίως ε, και την προηγούμενη θητεία κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι για τέτοια ζητήματα, κυρίως μετά τη Λισαβόνα, έτσι, δεν δε μπορούμε παρά να ε, το ως κοινοβούλιο όλα αυτά τώρα τα οποία συνδέονται με την ε, καλή κατάσταση των ζώων, κάνουμε μία ανοίξη, αλλά όσον αφορά το ζήτημα αυτό, υπάρχει μία εργασία σε βάθος και είναι σαφές ότι η καλή κατάσταση των ζώων ε, είναι άμεση προϋπόθεση για την ε, άριστη ποιότητα του προϊόντος. Και να σας πω και το εξής. Όταν εσείς παραγγέλνετε στο, στο, στο εστιατόριο ένα ψάρι, και ε, βλέπετε για παράδειγμα όταν ε, ε, βλέπετε την κατάσταση του ψαριού, βλέπετε τη σπονδυλική στήλη του ψαριού, άμα είναι στραβή καταλαβαίνετε ότι ήταν σε, ιδα, σε και υπέφερε. καταλαβαίνετε, πέραν δηλαδή της γεύσης, αυτό έχει να κάνει και με την ποιότητα και καταλαβαίνετε ότι το συγκεκριμένο ζώο υπέφερε σε κακές συνθήκες. Αυτό το λέω εν αστείο, αλλά θέλω να σας πω ότι και αυτό το ζήτημα, αν το παρουσιάσουμε καλά προς τα έξω, στα πλαίσια δηλαδή μια σαφού πολιτική ε, σήματο και πρόθεση του ευρωπαϊκού προϊόντο, τότε αποτελεί ένα παραπάνω πλεονέκτημα. Είναι κάτι το οποίο αγγίζει τον καταναλωτή. Το ξαναλέω και κλείνω εδώ. Η προσέγγιση που θα πρέπει να έχουμε και σε αυτή τη φάση Τροπολογία του εγγράφου είναι η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι εμεί σήμερα δεν γράφουμε τον κανονισμό. Διαφορετικά, το ξαναλέω, δεν θα αρκούσε. Θα ήταν ανεπαρκή αυτή η γνωμοδότηση. Αλλά και από στρατηγική άποψη. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να επισέλθουμε σε ιδιαίτερε λεπτομέρειε όσον αφορά την ουσία. Κοιτάξτε, βεβαίω, να διευκρινίσουμε τα πράγματα και να λάβουμε υπόψη τι παρατηρήσει των συναδέλφων. Αλλά αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να υπάρχει όσο εδώ περισσότερη συνένεση μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβουλίου για να ξεκινήσουμε αυτή την ε, πορεία. Εάν λοιπόν είναι θετική η άποψη ε, της και της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, τότε θα οδηγηθούμε τελικά στον κανονισμό και τότε θα ξεκινήσουμε πολύ συγκεκριμένα ε, την εργασία επί των λεπτομεριών και σίγουρα θα εντοπίσουμε αυτές τις ε, μικρές αντιφάσεις που με μια επιφανειακή ανάγνωση δεν ε, προκύπτουν. Και το ξαναλέω και τελειώνω. Υπάρχουν πράγματα που έχουν να κάνουν με το Ταμείο, για παράδειγμα, που ανέφερε η, Πρόεδρος Πρόεδρο, θέματα τα οποία αφορούν την ε, κοινή ελευθερική πολιτική. Και εγώ δεν αποκλείω και την περίπτωση αυτό το τμήμα, όταν θα γίνει νόμος πλέον, κανονισμός και όχι ε, ανακοίνωση να αποτελεί μέρος της κοινή ελευθερικής πολιτικής. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για κάτι ξεχωριστό. Ακριβώς γιατί υπάρχει αλληλεπίδραση και το είπα και προηγουμένως. Ανάμεσα στην εξέλιξη ή στη μη εξέλιξη της αλίας και στην, ε, και στην εξέλιξη της είναι άμεση λοιπόν η σχέση. Δεν είναι δύο ξεχωριστοί δρόμοι. Ίσως το πολύ να είναι παράλληλοι οι δρόμοι αυτοί, αλλά σίγουρα συνδέονται στενά. Σαν τις ράγες του τρένου. Παράλληλες, αλλά κοιτάξτε, ε, υπάρχει κάτι που ενώνει αυτές τις δύο παράλληλες ράγες του τρένου. Ευχαριστώ. Eh, λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Μιλάνα. «13 Απριλίου ε, στις 12 η ώρα ε, προθεσμία για τις ε, τροπολογίε. Και στι 4 Μαου, όπω είπε ο κ. Μιλάνο, θα ψηφίσουμε. Και τώρα πάμε στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξη που αφορά τι συγκεκριμένε τροπολογίες τη σύμβαση για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία ε, ΝΑΦΟ, όπω είναι γνωστό. Στην ε, τελευταία συνεδρία των συντονιστών μοιράστηκε η η έκθεση αυτή την πήρε το ΕΛΚ, δεν έχει οριστεί ακόμα εισηγητή, αλλά ε, θα προχωρήσουμε όμω την παρουσίαση τη πρόταση εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρόλο που έχουν έτσι τα πράγματα. Η κυρία Νίλσεν έχει το λόγο. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια ανακοίνωση σε μια απόφαση του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την έγκριση αυτών των τροπολογιών της Σύμβασης ε, ΝΑΦΟ. Είναι, πρόκειται για το έγγραφο της Επιτροπής 2010-75 τελικό φάνα. Οι ορισμένες τροπολογίε τροπολογίες αυτές είχαν ήδη εγκριθεί στην αγγλική τους εκδοχή από το 2007 και αργότερα μετά και στην γαλλική έκδοχη, οι τροπολογίες αυτές περιλαμβάνουν μια πολύ λεπτομερή ε, αναθεώρηση της ε, σύμβασης. Αλλά το βασικό άρθρο της σύμβασης παραμένει σε ισχύ. Το πρώην δηλαδή ε, άρθρο 22 το οποίο έχει λάβει τώρα τον αριθμό 23. Ε, πρόκειται δηλαδή για μια σχεδόν πλήρη αναθεώρηση της σύμβασης αφού μόνο και το άρθρο έχει μείνει έχει και ο ε, στόχος και οι βασικές αρχές της σύμβασης έχουν αναθεωρηθεί προκειμένου να ευθυγραμμίζεται πλέον η σύμβαση με πιο σύγχρονους τρόπους διαχείρισης της αλληλείας ειδικότερα λαμβανωμένες υπόψεις ε, της ε, έναξης ισχύω ε, της φωνή τη Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την διαχείριση των αποθεμάτων. Επίσης λαμβάνονται υπόψη στόχοι όπως η διασφάλιση των οικοσυστημάτων, των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, η συμμόρφωση με αντίστοιχη πολιτική, η ανάγκη διασφάλιση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και ούτω καθεξής. Επίσης έγιναν και κάποιες, αν θέλετε, διοικητικού χαρακτήρα ε, τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της ΝΑΦΟ. Έχουν δηλαδή ε, απλουστευτεί περισσότερο οι σχετικέ διαδικασίες. Έχουμε συγχώνευση μάλιστα το Προεδρείο και Γραμματέας. Ταυτόχρονα η... έχει εξυγχρονιστεί ο τρόπος ε, με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των υποθέσεων. Ο τρόπος λήψης ε, των αποφάσεων έχει επίσης βελτιωθεί και υπάρχει και μια νέα διαδικασία επίλυσης διαφορών. Η πρότασή μας λοιπόν είναι να εγκριθούν οι εν λόγω τροπολογίες της σύμβασης και είμαστε στη διάθεσή σας για να διευκρινίσουμε τυχόν σημεία που αφαιρούν αυτή την ε, πρόταση για την αγγλική Έχετε κάποια ερώτηση? Όχι. Επομένως, το κείμενο μας καλύπτει και έχουμε και τη δεδομένη νομική βάση που νομίζω ότι είναι η πιο σωστή. Εκτός αν προκύψει κάτι από τον μελλοντικό εισηγητή. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα πέραν αυτών. Ευχαριστούμε κύριε Νίλσα. Οι συντονιστές μας είναι εδώ. Α, όχι, όχι. Έφυγε, έφυγε μια συνάδελφος. Bueno, les pido a los coordinadores que a posible se queden y vamos... Οπότε, ας κάτσουν εδώ οι συντονιστές για να κάνουμε τη συνέντευξη τώρα αμέσω, χωρίς να κάτσουμε και να περιμένουμε μέχρι τις 8 η ώρα όπως προβλέπετε μπορούν να αποχωρήσουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι γιατί θα γίνει με κλεισμένο θυρών η συνεδρίαση.